So dear καλώς ήρθατε. Ενώ θα εγκρίνω την ημερήσια διάταξη, θα κάνω και μια σύντομη ανακοίνωση. Ένα διορθωτικό. Για την οδηγία 2013-36 του 2013 για τη μη πρόσβαση των θεσμών CRD4 μετά την διόρθωση από του νομικούς γλωσσομαθείς, κυκλοφόρησε στις 7 Δεκεμβρίου βάσει του άρθρου 231 του ιστορικού κανονισμού και αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις από την Επιτροπή, το διορθωτικό θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο. Θα ανακοινωθεί στην επόμενη Ολομέλεια ε, ή δυνατόν, μάλλον στην ε, Δεκεμβριανή και θα εγκριθεί εφόσον εάν ε, κάποια πολιτική ομάδα 40 μέλη με υπογραφές ζητήσουν να ψηφιστεί. Τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στο οικονομικό θέμα, στο διάλογο και την αντιλογή απόψεων με την Επιτροπή σχέδιο προπολογισμού, σχέδιο προπολογισμού για τα κάτι μέλη της Ευρωζώνης με τον ε, Επίτροπο Ντομπρόφσκης και τον Επίτροπο Μοσχοβησή. Καλώς ήρθατε, έχουμε αργήσει λιγάκι, οπότε αμέσως θα δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστούμε για την δυνατότητα να συζητηθούν ε, οι γνωμοδοτήσεις και οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τα κράτη-μέλη και την Ευρωζώνη. Από το 2008 μέχρι την εισαγωγή 2013 αυτού του εγχειρήματος που αποτελεί χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής ε, διακυβέρνησης για τον συντονισμό των πολιτικών μας δίνει μια ευκαιρία ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γνωμοδοτήσει σε σχέση με το σχέδιο προϋπολογισμού των κρατών μελών που στη συνέχεια ακολουθεί την κανονική διεργασία. Επίση, τα Εθνικά Κοινοβούλια μπορούν να, να γνωρίζουν σε βάθο το τι συμβαίνει σε σχέση με τις πολιτικές των άλλων κρατών μελών της ζώνης ευρώ. Επίση βοηθά τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν τα στοιχεία της ε, δημοσιονομική εξέλιξη. Έτσι λοιπόν σε σχέση με την συζήτηση αυτών των ε, γνωμών και την δημοσίευση τους που ολοκληρώνεται με τις ε, γνώμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις επιδόσεις ε, δημοσιονομικά των κρατών μελών. Μέσα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης οικονομικής συγκυρίας που ήδη προηγούμενα σε άλλες ακροάσεις έχουν αναφερθεί, εδώ θα τονίσω ένα κύριο στοιχείο εργαζόμαστε όσον αφορά μια μετριοπαθή οικονομική ανάπτυξη όμως όλα τα κράτη-μέλη αναμένεται να σημειώσουν ένα ποσοστό ανάπτυξης, ενδυναμώνεται η δημιουργία θέσεων απασχόλησης ε, όσον αφορά την ανάπτυξη και φέτος θα είναι πιο αυξημένο αυτό το ποσοστό από την έναρξη της κρίσης, όμως ταυτόχρονα αυτή η ανάκαμψη είναι ευάλωτη. Υπάρχει και πολιτική αβεβαιότητα, βραδείς οικονομική ρυθμή ανάπτυξης και υπάρχουν πολλές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Υπάρχει ακόμα υψηλό επίπεδο ανεργίας και υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα όσον αφορά τα, τα ποσοστά ανάπτυξης, τα ποσοστά υπερχρέωσης καθώς επίσης και τις προοπτικές και την δημιουργία βελτιωμένου κλίματος στα κράτη-μέλη όσον αφορά την ανάπτυξη δεδομένου αυτού του σκηνικού αξιολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν η δράση των κρατών μελών ευθυγραμμίζεται με τους κοινού κανόνες και την συμμετοχή τους στην κοινή προσπάθεια στην Ευρωζώνη. Ποια εικόνα είναι αυτή που απορρέει συνολικά για τα κράτη-μέλη. Πρώτα λοιπόν πρέπει να σημειώσουμε ότι όσον αφορά τα ελλείμματα θα συνεχίσουν να μειώνονται για να φτάσουν το 1,5% σε σχέση με το 1,8% που είχαμε φέτος και 1,9 ε, πέρυσι. Επίσης ε, το μέσος όρος ε, χρέους μειώνεται και αυτός ενώ είχε φτάσει στην κορυφή στο στέγα, στο αποκορύφωμά του το ε, ε πέρσι και τώρα συνεχίζει να μειώνεται σταδιακά. Και είναι αξιοπρόσεκτο ότι του χρόνου μόνο ένα κράτος μέλος της Ευρωζώνης θα εξακολουθεί να έχει ένα ε, έλλειμμα πάνω από 3% του ΑΕΠ. Έτσι λοιπόν αν αξιολογήσουμε τα, την ευθυγράμμιση των κρατών μελών όσον αφορά τα, τα σχέδια προϋπολογισμού που έχουν ε, καταθέσει θα δούμε ότι σε μεγάλο ποσοστό είναι ουδέτερο αυτό το πλαίσιο κατά το 2017 και όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις της πρότεινε μια μετριοπαθή ε, πολιτική επέκτασης ε, αξίζει να σημειώσουμε ότι βρισκόμαστε μέσα σε μια ιδιαίτερη συγκυρία όπου οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής πολιτικής ε, θεωρείται ότι είναι πιο ε, αποτελεσματικές οι δράσεις μέσω της ε, δυνατότητας μόχλευσης όσον αφορά την νομισματική πολιτική δεν σημαίνει αυτό ότι θα ε, πρέπει να αγνοηθεί ο συντονισμός και πρέπει να δημιουργηθούν οι δυνατότητες ώστε να μπορέσει η συλλογική αυτή προσέγγιση να αποδώσει καρπούς. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι υπάρχει περιθώριο να βελτιωθεί η ποιότητα των δημοσιονομικών όσον αφορά τις ε, επενδύσεις, ε, τις διαφορετικές ε, μεταρρυθμίσεις και την αποτελεσματικότητα. Και έτσι όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές η αξιολόγησή μας πρέπει να είναι διαφοροποιημένη σε σχέση με τα κράτη-μέλη ανάλογα με τα ποσοστά που επιτυγχάνονται κράτη-μέλη με υψηλό ποσοστό ε, χρέους ε, πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση και να υπάρχουν και οι ρήτρες ευελιξίες ε, κράτη τα οποία έχουν υπερβολική, υπερβολικό χρέος πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους με τις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις. Υπάρχει όμως ένα, μια ομάδα κρατών μελών που πρέπει να δημιουργήσει επαρκή επαρκή περιθώρια για επενδύσεις ώστε να δημιουργηθούν προοπτικές ανάπτυξης ε, να αντιμετωπιστούν ε, τα προβλήματα των χωρών που αντιμετωπίζουν τέτοιες προκλήσεις. Ε, επίσης, τα κράτη-μέλη τα οποία πρέπει να παροτριθούν και να ενθαρρυνθούν να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις τους και εδώ θα γίνει περισσότερο λόγος για συγκεκριμένες τοποθετήσεις για συγκεκριμένες χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μας καλέσατε για τέταρτη φορά για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Από την εισαγωγή του ΤΟΥΠΑΚ γίνονται αυτές οι ανταλλαγές. Αυτός ο διάλογος βασίζεται στο ΤΟΥΠΑΚ και είναι πολύ σημαντικός για τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης και ενισχύει αυτό που επιθυμούμε, τη διαφάνεια της ε, διαδικασίας. Ε, μπορώ να σας παρουσιάσω διάφορα έγγραφα που δημοσίευσε στις 16 Νοεμβρίου Κομισιόν στα πλαίσια του πακέτου για το φθινόπωρο του 2017 και έχουν την ανακοίνωση για έναν θετικό προσανατολισμό της δημοσιονομικής πολιτικής Ευρωζώνης που μόλις σας παρουσίασε ο Βαλδής, μια βασική ανακοίνωση με οριζόντια συμπεράσματα για τα δημοσιονομικά σχέδια της Ευρωζώνης, 18 γνωμοδοτήσεις για τα ε, σχέδια. Η Ελλάδα είναι υποπρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής και έχει μια άλλη διαδικασία. Η Ισπανία και η Λιθουανία έστειλαν τα δημοσιονομικά σχέδια ε, που είναι για... με απαράλλακτη πολιτική λόγω υπηρεσιακής κυβέρνηση τη στιγμή της παρουσίασης των σχεδίων. Σύμφωνα με τις διατάξεις λοιπόν του Συμφώνου και Ανάπτυξης, αυτές οι δύο χώρες θα πρέπει να στείλουν τα επικαιροποιημένα δημοσιονομικά σχέδια μόλις αποκτήσουν απόλυτη δημοσιονομική εξουσία οι νέες κυβερνήσεις. Ε, και η Ισπανία το έκανε την περασμένη Παρασκευή. Δύο ανακοινώσει για τη δράση της τη Ισπανική στα, στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, Η Κομισιόν έφτασε στο συμπέρασμα ότι και η Ισπανία και η Πορτογαλία πήραν τα απαραίτητα δημοσιονομικά μέτρα για την ε, χρονιά 2016 και επομένως δεν υπάρχει λόγος να αναστείλουμε τη χρήση των διαφορετικών ταμείων και επενδυτικών ταμείων. Επομένως η Κομισιόν, και αυτό είναι συμπέρασμα, ε, συνέχεια και του διαλόγου που είχατε μαζί, δεν πρότεινε την αναστολή για την Ισπανία και την Πορτογαλία. Τώρα, τα βασικά μηνύματα του πακέτου του 2017 είναι τα εξή. Ε, Όπω είπε ο Βαλτή, για πρώτη φορά η Κομισιόν καθόρισε το προσανατολισμό τη μεσονομική πολιτική για την Ευρωζώνη. Είναι πολύ σημαντικό για την εμβάθυνση τη ΟΝΕ σε ό,τι αφορά τις επιμέρους χώρες, να σας πω ότι οι στόχοι μας είναι οι εξή. Αυτοί που έχουν δημοσιονομικό περιθώριο θα πρέπει να ξοδεύουν περισσότερο και να επενδύουν περισσότερο, ενώ αυτοί που, είναι, που υπολείπονται σε σχέση με τους στόχους θα πρέπει να επικεντρωθούν στις δημοσιονομικές τους δεσμεύσεις. Οι υποχρεώσεις του συμφώνου είναι διτές για τα κράτη-μέλη ανάλογα με την δημοσιονομική τους κατάσταση. Και αυτό είναι το μήνυμα που δείχνουν, ε, που δείχνουν ε, οι 18 μας νομοθετήσεις. Ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε την αυστηρή εφαρμογή, αλλά έξυπνη εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, να σεβαστούμε τους κανόνες, ε, χρησιμοποιώντας την ευελιξία εκεί που προβλέπεται. Εκεί έχουμε φτάσει. Για τα κράτη-μέλη, που το ονομαστικό έλλειμμα είναι κάτω του 3%, δηλαδή στο προληπτικό σκέλος του συμφώνου, αξιολογούμε τον κίνδυνο απόκληση σε σχέση με αυτό που ονομάζουμε τον στόχο τον ενδιάμεσο Medium Term Objective, MTO, ε, ή την απόκληση σε σχέση με την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν για αυτό το στόχο. Τα κράτη-μέλη που το ονομαστικό τους ε, έλλειμμα είναι ανώτερο του διορθωτικό κλειδός του συμφώνου, ο κίνδυνος μη συμμόρφωση αξιολογείται με βάση τη ε, σύσταση του Συμβουλίου, με βάση το άρθρο 126.7 της συνθήκης, για να επανέλθει στο κατόφλι του 3% και να περάσουν στο προληπτικό σκέλος του, του συμφώνου. Πέρυσι κανένα κράτος μέλος δεν ήταν αντικείμενο μη συμμόρφωση ιδιαίτερα σοβαρή. Επομένω, η Κομισιόν δεν ζήτησε ε, σε καμία περίπτωση ένα θεωρημένο προπολογισμό από κανένα κράτο μέλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα πάνε καλά. Ε, η αξιολόγηση μα δείχνει ότι υπάρχουν διάφοροι βαθμοί κινδύνου και ζητάμε εκεί που είναι απαραίτητο να ληφθούν απαραίτητα μέτρα από τα κράτη-μέλη, ώστε να εξασφαλιστεί ο σεβασμό των κανόνων του Συμφώνου ε, Σταθερότητα Ανάπτυξη. Για τα κριτήρια που σα ανέφερα, την αξιολόγηση των κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη που είναι στο προοπτικό σκέλος. Υπάρχουν πέντε χώρες που ε, σέβονται το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Η Γερμανία, Εστονία, Λουξεμβούργο, Σλοβακία, κάτω χώρε. Τρει από αυτέ τι πέντε χώρε, η Γερμανία, οι κάτω χώρε και το Λουξεμβούργο, είναι πάνω από τον ενδιάμεσο ε, στόχο και ενθαρρύναμε τις χώρες αυτές να χρησιμοποιήσουν το δημοσιονομικό τους περιθώριο για να αυξήσουν τις επενδύσεις, διατηρώντας όμως τη διατηρησιμότητα των δημοσίων οικονομικών τους μακροπρόθεσμα. Τέσσερις χώρες είναι γενικά σύμμορφες με το σύμφωνο, Ιρλανδία, Λετωνία, Μάλτα και Αυστρία. Σε αυτήν την περίπτωση η απόκληση από τον ενδιάμεσο στόχο είναι κατώτερη από το 0,5 του ΑΕΠ και αυτή η απόκληση είναι ιδιαίτερα ασθενή στην περίπτωση της Λετωνίας. Αυτές οι χώρες σέβονται τον κανόνα του χρέους. Το χρέος της Λετωνίας είναι 40% του ΑΕΠ το 2016. Και προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να μειώνεται, ενώ το χρέος της Μάλτας θα μειωθεί και θα κατέβει κάτω από το όριο αναφορά στο 60% του ΑΕΠ το 2017. Στην περίπτωση τη Αυστρία η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη την επίπτωση του επιπλέον κόστου που συνδέεται με του πρόσφυγες, σε ό,τι αφορά την Ιρλανδία. Ένα σημαντικό τμήμα των ε, εσόδων από το εταιρικό φόρο χρησιμοποιήθηκε για να χρηματοδοτηθούν επιπλέον δαπάνε το 2016. Αυτό είναι αντίθετο στι ειδικέ συστάσει αναχώρα που ενθαρρύνουν την Ιρλανδία να χρησιμοποιήσει αυτά τα κέρδη, ούτω ώστε να επιταχύνει την μείωση του ελλείμματο και του χρέου. Έξι κράτη-μέλη ε, από την σκοπιά τη πρόληψη ε, παρουσιάζουν μη συμμόρφωση με το σύμφωνο. Τα, τα κράτη-μέλη αυτά κλήθηκαν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθούν με όσα προβλέπει το σύμφωνο. Είναι το Βέλγιο, η Ιταλία, η Κύπρο, η Λιθουανία, η Σλοβενία και η Φιλανδία. Σε ό,τι αφορά την Ιταλία, Έχουμε παρατείνει την περίοδο εφαρμογή τη ρήτρα που έχει να κάνει με του πρόσφυγε από το 2007. Μία ρήτρα που έπρεπε να ισχύσει μόνο για το 2015 και 2016 αρχικά. Γιατί το κάναμε αυτό, δεδομένη τη ένταση και τη αιμονή του μεταναστευτικού φαινομένου. Έτσι ακολουθήσαμε αυτό που μας κάλεσε να κάνουμε τον Οκτώβριο τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια με την σημαντική συμβολή, συμπεριλαμβανομένη τη οικονομική συμβολή, από κάποια κάτι μέλη που βρίσκονται στην προστοφυλακή τα τελευταία χρόνια. Θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι πρόσθετα, ε, προσωρινά μάλλον, για τα πρόσθετα κόστη που είχε να αναλάβει η Ιταλία, ιδίω με τα σεισμικά φαινόμενα, που είναι και συστηματικά και συχνά και μεγάλων διαστάσεων στην Ιταλία. Αυτό δεν είχε καμία βέβαια επίπτωση στην τελική αξιολόγηση του δημοσιονομικού σχεδίου της Ιταλίας που κινδυνεύει με τιμή συμμόρφωση ό,τι αφορά την Φιλανδία και την Λιθουανία. Κλήθηκαν ε, να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα για τις διευθυντικές μεταρρυθμίσεις, ιδίω η Φινλανδία τη ρήτρα για τις ε, για τι διοικητικέ μεταρρυθμίσει και η Φινλανδία κλείθηκε να περάσει σε επενδύσει. Αυτά θα αξιολογηθούν την άνοιξη. Ούτε αφορά το διευθυντικό σκέλο. Η Γαλλία γενικώ είναι σύμφωνοι με τους κανόνες του συμφώνου, ενώ η Ισπανία και η Πορτογαλία μπορεί και να βρεθούν σε μη συμμόρφωση. Η Γαλλία χρειάζεται διόρθωση του ελλείμματος εντό των πλαισίων των προβλέψεών μα, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική προσπάθεια και όχι χαμηλότερη από αυτή που είχε συσταθεί. Αυτό ελπίζουμε ότι μπορεί να βελτιωθεί αν δεν αλλάξουν τα πράγματα το 2018. Όμως, έχει και το ποσοστό 3,1% να αντιμετωπίσει η Γαλλία το 2018. Είναι μεγάλες προσπάθειες ακόμη και για το ελάχιστο αποτέλεσμα. Σε ό,τι αφορά την Ισπανία, θα εξετάσουμε και πάλι το εγχώριο καθάριστο προϊόν την ερχόμενη Παρασκευή με τη συμμετοχή των Ισπανών. Ακόμη δύο λόγια για τι επόμενε φάσει. Πρώτα απ' όλα περιμένουμε ένα δημοσιονομικό σχέδιο το οποίο να είναι επικαιροποιημένο από τι λιθουανικέ αρχέ, Θα κάνουμε την αξιολόγηση αυτών των σχεδίων μόλι μπορέσουμε. Δεν έχουμε ακόμη υποβάλει νέε εκθέσει βάσει του άρθρου 126.3 τη συνθήκη για τι χώρε που δεν τον κανόνα του χρέους, ιδίω την Βέλγια και την Ιταλία. Και περιμένουμε την ολοκλήρωση των προπολογισμών των χωρών αυτών για να υποβάλουμε τι εκθέσει ε, αμέσω μετά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, αυτέ ήταν οι συγχωρικέ μου παρατηρήσει για τη δέσμη μέτρων του φθινοπόρου 2017. <clears throat> Πέραν των όσων είπε ο Βάλτη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και πρώτος ο κύριος Μπάλτς από σού θα παρέμβουν. Ευχαριστώ θερμά κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σχετικά σύντομος, μια και έχει προχωρήσει ο χρόνος. Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο κύριο Ντομπρόφσης και τον Επίτροπο Μοσκοβισή θερμά για τα όσα μας εξέθεσαν. Με ενδιαφέρει ένα ζήτημα ιδιαίτερα. Και επ' αυτού απόψε θέλω να διατυπώσω μια ερώτηση. Τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν σαφώς πιο αισιόδοξε προοπτικές όσον αφορά την αύξηση, την ανάπτυξή τους και όσον αφορά το έλλειμμά τους και το διαθωτικό τους έλλειμμα σε σχέση με τις προοπτικές που διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις Γερμανία, Ολλανδία, Εσθονία, Μάλτα. Η ερώτησή μου τώρα επικεντρώνεται στο εξή ε, θέμα. Για ποιο λόγο τα περισσότερα κράτη-μέλη στην ε, αλληλεγγύη και στην ε, ισχύ τους φαίνεται να υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους. Γιατί συμβαίνει αυτό. Μια άλλη ερώτηση. Με με υπερβολικά αριθμητικά μεγέθη καταλήγουν σε συσκέψεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μπορέσουν τα μέγιστα να επιτύχουν και να είναι υποχρεώσεις τους οι ελάχιστες δυνατές. Γιατί συμβαίνει αυτό. Ευχαριστώ. Απάντηση. Λοιπόν, πολύ καλά. Σε αυτό το ερώτημα πράγματι συμβαίνει ότι οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι προβλέψεις για τις προοπτικές των κρατών μελών διαφέρουν δεν είναι πάντα ακριβώς οι ίδιες. Ωραία. Και πρέπει να πούμε ότι δεν είναι τίποτα το δραματικό όμως σε σχέση με αυτές τις παρεκκλήσεις, αλλά πολλές φορές οδηγούν σε διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις προοπτικές και τα σενάρια, όσον αφορά την δική μας αξιολόγηση που περιορίζονται σε κάποιες ποσοστιαίες μονάδες ή σε κάποια δεκαδικά των ποσοστιαίων μονάδων. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, όταν αξιολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη συμμόρφωση των κρατών μελών όσον αφορά τους όρους ε, του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, λαμβάνει πάντα υπόψη τις ε, προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά κανόνα. Πρώτα, αξιολογείται αν τα ίδια τα κράτη-μέλη στοχεύουν να συμμορφωθούν ...για να ανταποκριθούν με τις συστάσεις ε, του Συμβουλίου για να ανταποκριθούν ε, στους δημοσιονομικούς στόχους. Αυτό μετράται και αξιολογείται πρώτον και επίσης ε, γι' αυτό αξιολογούμε αν υπάρχει ίσως σοβαρή μη συμμόρφωση. Σε σχέση με τις γνωμοδοτήσεις μας στη συνέχεια λαμβάνουμε υπόψη τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως βάση για αυτή τη διαδικασία αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν ε, τα κράτη-μέλη με υπερβολικά αισιόδοξε εκτιμήσεις ε, να δίνουν μια διαφορετική εικόνα της κατάστασης που βελτιώνει τα πράγματα σε σχέση με την πραγματική εικόνα. Ευχαριστώ. Για την παρατήρηση του κ. Μπάλτς, δίκιο έχετε. Όμως, κάναμε πολλή προσπάθεια και για να δούμε αν εφαρμόζονται σωστά οι κανόνε του συμφώνου. Τώρα, όπως είπε και ο Βάλτη, βλέπει το Συμβουλίο ότι οι αποκλήσει είναι ελάχιστε. Υπάρχει λοιπόν πρόεδρο ω προ ως τη διαδικασία σύγκληση, ιδίω. με την προστασία των ιδιωτών. Τώρα οι μεθοδολογίε που χρησιμοποιούμε είναι αυτέ που κρίναμε καταλληλότερες και είναι ίδιε για όλου. Ε, ασχέτως του ποια είναι η χώρα ή η φάση του πολιτικού κύκλου. Ο πολιτικό ε, κύκλο, το σημείο του κύκλου μπορεί να παίξει ρόλο. Το 2017 θα είναι μια χρονιά πλούσια εκλογέ. Όμω, αυτό δεν σημαίνει ότι στο τέλο δεν μπορούμε να πετύχουμε τη μείωση τη ψαλίδα, την κάλυψη τη ψαλίδα για πολλά θέματα που μα απασχολούν. Ευχαριστούμε, κυρία Μπερέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Το είπατε πολύ καλά και το περιγράψατε με λεπτομέρειες. Οι χώρες βγαίνουν τώρα λίγο από φουρτούνα. Κανείς δεν βρίσκεται στην ακρίβεια των κανόνων του Συμφώνου και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αυτό μας αφήνει κάποιο περιθώριο ελιγμού για να ξαναδούμε τα στοιχεία της διάγνωσης. Ε, μήπως στη δική σας αξιολόγηση των ε, δημοσιονομικών προγραμμάτων, των ετήσιων προπολογισμών φτάσατε στα όρια των όσων μπορούσατε να κάνετε. Έχω και μια δεύτερη ερώτηση, διότι ξεκινήσατε μια σημαντική συζήτηση με τις συστάσεις σας για την Ευρωζώνη και τη σχετική ανακοίνωση για, την, ε, για το δημοσιονομικό προσανατολισμό. Είναι κάτι που το ζητούσαμε εδώ και πολύ καιρό. Πώς όμως ε, αυτή αυτός ο συναθρισμένος δημοσιονομικός ε, προσανατολισμός θα πάρει διαφορετική έκφανση στην περίπτωση του κάθε κράτους μέλους. Αυτή η συνάθρηση του δημοσιονομικού προσανατολισμό, εφόσον τώρα βγαίνουμε από την καταιγίδα, από τον κυκλώνα, μπορεί να πάει λίγο πιο μακριά και να ανοίξει η συζήτηση για ένα είδος ε, χρυσού κανόνα, του χρυσού μισθού και του σχετικού κανόνα, δηλαδή να προβλέψουμε μήπως είναι ελάχιστο μισθό για τα κράτη της Ευρωζώνης. Και τέλος, θα μου πείτε, είναι πολύ νωρίς για να το πούμε τώρα αυτό, αλλά παρόλα αυτά θα το πω, θέλω να ρωτήσω και για τη συνεισφορά του European Fiscal Board διότι για πρώτη φορά είδαμε να παρεμβαίνει στην όλη συζήτηση. Πώς αξιολογείται αυτή την παρέμβαση και τι να αποκομίσουμε κι εμείς από τη δική σας την ε, κρίση για να το χρησιμοποιήσουμε στην επόμενη συζήτηση μαζί τους. Ωραία. Πρώτα, για την ε, διάγνωση και το αν υπάρχει περιθώριο ελιγμού. Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ η οικονομική ανάκαμψη συνεχίζεται, προσκρούει σε αβεβαιότητες και ασάφειες από την προηγούμενη κατάσταση, οπότε δεν υπάρχει περιθώριο για αυταρέσκεια. Ε, πρέπει να αποφασίσουμε στο ευρωπαϊκό εξάμενο αν θέλουμε να επικεντρωθούμε στις επενδύσεις, στις σοβαρές δημοσιονομικές πολιτικές, την πολιτική επασχόληση ή αν θα κοιτάξουμε τις ανισότητες στο εισόδημα και την συμμετοχική άνοιξη ενδεχομένως. Αυτό πιστεύω ότι το χρειάζεται απελπιστικά ο κόσμος. θέλουν οι μικρονομικοί όροι και αριθμοί που χρησιμοποιούμε να φέρουν και χειροπιαστά αποτελέσματα για όλους. Αυτό θα φανεί και στις ανασύσταση, στις αναχώρασεις τάσεις μας μάλλον, όταν θα ασχοληθούμε και σε επίπεδο άλλων πολιτικών με τη μείωση των διαφορών στο εισόδημα. Μετά θίξατε το θέμα των των μισθών και τα λοιπά. Θα έλεγα ότι αυτά μπορεί να καλυφθούν από τον λεγόμενο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα, ο οποίος αυτή τη στιγμή χτίζεται και ο οποίος ελπίζουμε θα καλύπτει τις κοινωνικές προεκτάσεις και ζητήματα που μας απασχολούν για το θέμα του European Fiscal Board και πώς ε, το βλέπουμε εμείς. Ε, το πρόβλημα δεν είναι θεσμικό, διότι το Fiscal Board στόχο είχε να αξιολογήσει την Επιτροπή και τις αναλύσεις της, όχι αντιστροφώς. Μην αρχίσουμε τώρα να αξιολογούμε εκείνους που μας αξιολογήσανε. Καλό θα ήταν να σεβαστούμε το θέμα πώς διοργανώθηκε. Αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο και πρέπει να το σεβαστούμε. Το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Σώμα δημιουργήθηκε ως ανεξάρτητος φορέας και έτσι θα παραμείνει. Μάλλον είναι πολύ νωρίς για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Δύο λόγια να προσθέσω κι εγώ. Πρέπει να σεβαστούμε φυσικά την ε, ανεξαρτησία του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, του European Fiscal Board, αλλιώ θα ήταν και άκομψο και άτιμο εκ μέρου μας. Παρότι αυτός ο οργανισμός μόλις ξεκίνησε τις εργασίες του, πρέπει να σημειώσουμε ότι στις ε, συζητήσεις του Eurogroup ο πρόεδρος του παρενέβη και μίλησε όντα το ίδιο μήκο κύματο με εμά για το συνολικό δημοσιονομικό προσανατολισμό. Δηλαδή, ο πρόεδρος του European Fiscal Board και η Κομισιόν είχαν την ίδια άποψη. Και ακριβώς ο ρόλος του αυτός είναι, γιατί ε, στο θέμα αυτό και εμείς και εκείνοι δρούν προς το συλλογικό συμφέρον. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις. Πριν από λίγους μήνες, κάποιοι ε, συνάδελφοι υπέβαλαν γραπτές ερωτήσεις στην Κομισιόν και σας ρωτούσαμε για διευκρινήσεις για την ακριβή μεθοδολογία και την ανάλυση που χρησιμοποιείται για να καθοριστεί το αν ένα κράτος μέλος συμμορφούνται με την ρεσιμότητα της, δημοσιο... της δημοσιονομικής του βοήθεια. Η απάντηση ήταν πολύ αόριστη και χωρίς ουσία. Για εμάς ως μέλη της Επιτροπής ΕΚΟΝ είναι πολύ σημαντικό να ελέγχουμε τα, την οικονομική βοήθεια που μοιράζεται στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να ρωτήσω ξανά. Η Κομισιόν μπορεί να εξηγήσει πώς ακριβώς αξιολογεί τη συμμόρφωση με τα προγράμματα όταν χρησιμοποιεί ποια ανάλυση, ποια μεθοδο, για να το κάνει αυτό. Και η δεύτερη ερώτηση αφορά ένα διαφορετικό υπολογισμό. Ζητήσατε περισσότερες επενδύσεις από τα κρέα κράτη-μέλη τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο και τις κάτω χώρες που έχουν κάποιο δημοσιονομικό περιθώριο. Η ε, στατιστική υπηρεσία της Ολλανδίας υπολόγισε ότι αν αυτές οι τρεις χώρες, Γερμανία, Ολλανδία ε, και Λουξεμβούργο χρησιμοποιήσουν όλο το δημοσιονομικό περιθώριο που θα έχουν, θα είναι περίπου το 50% του 0,5% του ΑΕΠ που προτείνετε εσείς. Δηλαδή, πώς υπολογίσατε ότι 50 δισεκατομμύρια θα πρέπει να επενδυθούν επιπλέον. Με ποια μέθοδο φτάσατε σε αυτό το νούμερο. Ευχαριστώ. Uh, well, uh, on, on the first question. Για το πρώτο ερώτημα, για τη συμμόρφωση με τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής. Οι όροι υπάρχουν στο μνημόνιο που υπογράφει τον λόγο κράτος μέλος. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο ένα κράτος μέλος ε, υποπρόγραμμα που είναι η Ελλάδα. Επομένως υπάρχει ένα μνημόνιο όπου όλοι οι όροι και οι προποθέσει αναφέρονται και συνεχεία υιοθετείται από το Συμβούλιο το μνημόνιο αυτό. Και η Κομισιόν αξιολογεί τη συμμόρφωση σημείο προς σημείο. Κάποια στοιχεία, όπως παραδείγματο χάρη δημοσιονομικοί στόχοι, ας πούμε το πρωτογενές πλεόνασμα κτλ. Όλα αυτά τα μετράμε με νούμερα και κάνουμε την αξιολόγησή μας ε, και με βάση τις οικονομικές ε, προβλέψεις για την Ελλάδα. Υπάρχουν κάποια άλλα σημεία τα οποία είναι πιο ποιοτικά. Αξιολόγηση Φερρυπίν των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων και την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι διαφορετικέ μεταρρυθμίσει. Κάνουμε μια αξιολόγηση, αλλά ανασημείο, με βάση τα όσα προτείνει και όσα λέει ρητά το μνημόνιο. Μερικές φορές είναι λοιπόν η αξιολόγηση αυτή είναι ποσοτική, άλλες φορές είναι ποιοτική, για να δούμε αν συμμορφούνται η χώρα και σε ποιο βαθμό. Και πέρα από το μνημόνιο, για τις επόμενες ε, αξιολογήσεις έχουμε και τα λεγόμενα milestones, που είναι οι λεπτομέρειες των όσων πρέπει να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη. Η δεύτερη ερώτησή σας για το συνολικό δημοσιονομικό προσανατολισμό. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι η ανακοίνωση της Κομισιόν μιλούσε για ένα δημοσιονομικό προσανατολισμό μέχρι 0,5%. Δηλαδή θετικό δημοσιονομικό προσανατολισμό μεν, αλλά μέχρι το 0,5% του ΑΕΠ. Αυτό προέρχεται από μακροοικονομικές σκέψεις. Ένα δημοσιονομικό προσανατολισμό που θα μας επιτρέψει να κλείσουμε το μισό από το υπάρχον παραγωγικό κενό στην Ευρωζώνη. Φυσικά, απόκειται στα κράτη-μέλη να κάνουν διαβουλεύσεις κτλ. Γι' αυτό δεν βάζουμε κανένα νούμερο δίπλα σε αυτό το δημοσιονομικό προσανατολισμό. Δεν βάζουμε ποσό που το ή κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσουν σε αυτό το πλαίσιο. Ο Πιέχ, δεν ξέρω αν έχει να πει κάτι γι' αυτό. Το 0,5% θα είναι το μέγιστο και για μας δεν ήταν και το πιο σημαντικό πράγμα. Το πιο σημαντικό ήταν η, ότι η έννοια του δημοσιονομικού προσανατολισμού τέθηκε. Το fiscal stance τέθηκε. Ότι θα πρέπει να είναι, να είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αφορά όλη την Ευρωζώνη. Το δέχτηκαν όλοι. Και είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο όπου όλο και περισσότερε χώρε ε, έχουν περισσότερο δημοσιονομικό περιθώριο και ζητάμε να το χρησιμοποιήσουν. Το νούμερο δεν ήταν το πιο σημαντικό πράγμα λοιπόν. Κάποιοι υπολογισμοί Φτάνουμε, μέσα στο 0,25% και όχι στο 0,5%. Actually, το Μεταξύ 0,3 και του 0,8 ήταν. Έχει φτάσει στο 0,5 τώρα. Η Μαρίζα Ματίας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πριν απ' όλα, η η είδηση τη αναστολή των ιδιωτικών κονδυλίων είναι καλή είδηση. Το πρόβλημα είναι ότι υπήρξαν αμφιβολίε από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό έχει να κάνει με τι αμφιβολίε τη το θεσμικό οργάνο που, με το οποίο συζητάμε εδώ. Ήθελα λοιπόν να μιλήσω για το θέμα της δημοσιονομικής σταθερότητας που χρησιμοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως τη βόλευε και υπήρχε συγκεκριμένη περίπτωση της χώρας μου, της Πορτογαλίας. Η κυβέρνηση έλαβε τα καθήκοντά της και μια εβδομάδα μόλις μετά μας προέκυψε ένα καινούριο σκάνδαλο, σκάνδαλο δημοσίου χρήματος. Αυτό είχε να κάνει με φόρους και μέχρι με βιαστικές ιδιωτικοποίησεις. Σήμερα υπάρχει έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου που ε, σχολιάζει το πώς ε, προχώρησε η διαδικασία για, την, ε, για το Γενικό Ταμείο Καταθέσεων, δηλαδή την Εθνική Τράπεζα της Πορτογαλίας, και τις ε, διαδικής διευκολύνσεις που δίνονταν από εκεί. Από αυτή την τράπεζα ξεκινήσανε διευκολύνσεις για πολλές άλλες. Θα μπορούσα να κατονομάσω πολλές. Αυτό δημιούργησε φοβερές επιβαρύνσεις στον προπολογισμό μας και δημιούργησε φοβερή έλλειψη ισορροπίας. Διαφυγή. Ξέρετε, Επιτροπή, ποιες είναι οι αποφάσεις των ε, τεχνικών ομάδων που κρύβονται στα Υπουργεία των ε, κυβερνήσεων και των κρατών μελών και που πίσω από κλειστέ πόρτες μπορούν να κανονίσουν όλα αυτά τα, όλες αυτές τις αποφάσεις αλλά εμείς μετά αν δεν γίνονται αυτά δημόσια πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι δεν έχουν συνενοχή στην ε, υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος στην απόκρυψη και την κλοπή δημόσιου χρήματος αυτά καλύφθηκαν από κάποιους από ομάδες τεχνοκρατών που η Επιτροπή, εάν δεν τις έκανε κρυφά, ίσως ε, θα καταλάβαινε ότι το κοινό αυτό το ενδιαφέρει. Θα ήθελα να διευκρινίσω σε ποιο πλαίσιο ε, αναγκαστήκαμε να πιθανολογήσουμε την αναστολή των διευθυντικών κονδυλίων. Δεν ήταν τεχνοκρατική απόφαση για την κατανάλωση, την εκτέλεση των κοντιλίων, ε, την απόδοσή τους κτλ. Ήταν κάτι που είχε να κάνει με την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τι σκεφτήκαμε λοιπόν ότι έπρεπε να υπάρξουν διευκρινήσεις για τις επιστώσεις πληρωμών για το 2016. Για τις αναλήψεις μάλλον πιστώσεων. Ε, Πρώτα απ' όλα έπρεπε να σκεφτούμε πολύ σοβαρά να μπορούσαμε να ορίσουμε πρόστιμο. Είδε τον Ιούλιο, αποφασίσαμε ότι δεν θα υπάρξει πρόστιμο η κύρωση ούτε για την Ισπανία και για την Πορτογαλία, ούτε για την Πορτογαλία. Έπειτα ένα δεύτερο πράγμα που το προβλέπουν αυτομάτως οι κανόνε. Αν δεν υπάρξει σεβασμό των ε, δεσμεύσεων, τότε ε, πέρα από την πραγματική δράση, ανάληψη δράση, δηλαδή την κύρωση, μπορεί να υπάρξει αναστολή αναστολή των διευθυντικών κονδυλίων. Συζητήσαμε με του εκπροσώπου των ε, ενδιαφερομένων κυβερνήσεων, ε, Ισπανία, Πορτογαλία, και κανονίσαμε ένα διερθωμένο διάλογο με τη συμμετοχή τη Επιτροπή και εν τέλει όλε αυτέ οι προσπάθειε οδηγήθηκαν σε ένα κοινό αποτέλεσμα με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, ε, με τι αποφάσει των ηθινόντων τη Πορτογαλία και τη Ισπανία και βλέποντα ότι πραγματική δράση υπήρξε για το 2016 αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή αυτή μάλλον και μετά, η αναστολή για να καλυφθεί το πρόβλημα του δημοσίου δεν προτάθηκε. Το πρόβλημα δεν ήταν τα διορθωτικά κονδύλια, όπως είπα, ήταν οι αναλήψεις πιστώσεων πληρωμών από την Ισπανία και την Πορτογαλία. Από τη στιγμή που δεν τηρήθηκαν, εκεί σκεφτήκαμε να αναστείλουμε για να καλύψουμε. Ναι, αλλά η πραγματική ερώτηση που έθεσα για τις τεχνη... ομάδες τεχνοκρατών. Εκεί κάνουμε ό,τι μπορούμε για την αξιολόγηση. Η υπεύθυνη είναι η συνάδελφος Κρατσού. Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Δεν είπα ότι δεν υπήρχε ερώτηση. Είπα ότι δεν υπήρξε πρόβλημα που να δημιουργήσει θέμα αναστολής των διευθυντικών κονδυλίων. Ε, έληξε ο χρόνος. Εάν θέλετε ίσως γραπτός, διότι καταλαβαίνω ότι αναφέρεστε σε άλλο θέμα από ότι το πρόγραμμα αναφέρει. Εντάξει, θα το στείλω γραπτά, αλλά ε, η πραγματική ερώτηση δεν απαντήθηκε καθόλου. Σημειώνω ότι δεν δόθηκε απάντηση. Ο κύριος Γκίγκολ. Πρώτα θα ήθελα να πω το εξής. Καλωσορίζουμε την απόφασή σας για τα διαθροτικά ταμεία και είναι καλά μαντάτα αυτή η απόφασή σας. Είναι καλοδεχούμενη κίνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το δημοσιονομικό πρόγραμμα. Έχω μια ερώτηση κυριότερα. Το σκεπτικό για την απόφασή σας για την Ιταλία ποιο είναι αύξησε το έλλειμμα της η, Ιταλία. Ταυτόχρονα η Ιταλία αντιμετωπίζει την κατάσταση ότι κανονικά θα έπρεπε ο κανόνας για την υπερχρέωση να ισχύει, γιατί βρίσκεται επί αρκετό χρονικό διάστημα εκτός η e EDP. Όλοι γνωρίζουν ότι αν εφαρμοζόταν ο κανόνας για το χρέος θα μπορούσε να οδηγηθεί σε μια αποπληθωριστική κατάσταση και αυτό την επίδοση δημοσιονομικά της Ευρωζώνης θα την επιδίνωνε. Υπό το δικό μας πρίσμα. Όλα αυτά δεν δίνουν θετικό αποτέλεσμα. Δεν συνάδουν. Ταυτόχρονα μου δημιουργείται κάποια σύγχυση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή αξιολογεί ζητήματα που αφορούν την Ιταλία για να επι η προληπτική ανακεφαλαιοποίηση τουλάχιστον μια, μιας από τις τράπεζες της ενώ δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο και χώρος και ενώ υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως υπάρχει ανοιχτή πρόθεση για να λειτουργήσει αυτή η προληπτική ανακεφαλαιοποίηση για την κάλυψη απολειών σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό όμως αντιβαίνει το ε, πνεύμα των ε, συμπεφωνημένων Μπορείτε να μου εξηγήσετε ποιος είναι, ποιοι είναι οι κανόνες για την Τραπεζική Ένωση και τι συμβαίνει για τον κανόνα υπερχρέωσης όσον αφορά το δημοσιονομικό πακέτο μέτρων και πώς όλα αυτά συνάδουν στην περίπτωση της Ιταλίας. Δεν μπορώ να το κατανοήσω. Ποιο έγγραφο από εκατοντάδες σελίδες θα υπεξηγήσει όλα αυτά ώστε να μπορούν όλα αυτά να συνάδουν. Ευχαριστώ. Uh, Πρώτον, για την Ιταλία και τις δημοσιονομικές επιδόσεις της. Είναι κάτι που υπογραμμίζεται αυτό και στη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η, Ιταλία βρίσκεται στη διαχωριστική γραμμή της μη συμμόρφωσης και αυτό επίσης αντανακλάται στην αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη συμμόρφωση με τον κανόνα για την υπεχρέωση του, της Ιταλίας ε, για το 1.26 της, ε, της συνθήκης και αυτό αποτελεί στοιχείο το οποίο αξιολογείται όσον αφορά την ε, Ιταλία σε σχέση με, τη, με τα άλλα κράτη-μέλη όσον αφορά τις δημοσιονομικές επιδόσεις. Στη συνέχεια για τις καταστάσεις εκείνες στις οποίες κράτη-μέλη παρέχουν, προβλέπουν για παράδειγμα αδειοδότηση για τον τραπεζικό τομέα ή παρόμοιες δραστηριότητες από πλευράς τους έχουμε πολλά προηγούμενα κατά το παρελθόν όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι τέτοιου είδους ε, δαπάνες, τέτοιου είδους ε, δαπάνες τις αντιμετωπίζει ως ε, ένα ξεχωριστό πλαίσιο σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Και στη συνέχεια, όσον αφορά την σημερινή τρέχουσα κατάσταση, όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα στην Ιταλία, Πρώτα απ' όλα, όπως προηγούμενα ανέφερα στον προηγούμενο γύρο παρεμβάσεων, στον οικονομικό μας διάλογο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σχολιάζει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις το τι συμβαίνει με συγκεκριμένες τράπεζες. Ωστόσο, μέσω της δικής μας δράσης υπάρχουν διαφορετικές, διαφορετικοί τρόποι να αντιμετωπιστούν ε, ε, τραπεζικά ζητήματα και έναντι του ιδιωτικού τομέα την αναζήτηση δηλαδή λύσεων όσον αφορά και το πλαίσιο της ε, παροχής κρατικής επιχορήγησης ή βοήθειας. Μία αποσαφήνιση κατανόησα σωστά θεωρείται ότι θα πρέπει η προληπτική επανακεφαλαίωση και οι δαπάνες αυτές θα, εξαρτώ, θα θεωρείται ότι εντάσσονται στον κανόνα υπερχρέωσης. Για τον κανόνα αυτό ωστόσο θα διορθώσετε, θα προσαρμόσετε τα αριθμητικά μεγέθη όχι. Αυτό μου φαίνεται αξιοπρόσεκτο. Υπάρχει μια αλληλοδιασύνδεση εδώ σε σχέση με την ε, προληπτική ανακεφαλαίωση και το σύστημα, ε, το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Τι δηλαδή πρέπει να γίνει και πώς εντάσσονται τα κράτη σε σχέση με το προληπτικό σκέλος και το διορθωτικό σκέλος σε σχέση με τον κανόνα αυτό, διότι πρέπει να συνάδουν τα μέτρα αυτά και όταν αξιολογούμε εμείς από πλευράς μας ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία τα οποία οδηγούν σε παρέκκληση πρέπει να συνάδει ο τρόπος ε, της αξιολόγησης και των μέτρων ε, συμμόρφωσης ε, όσον αφορά την τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των κανόνων και κανονισμών που έχουμε θεσπίσει και αυτά πρέπει να αξιολογηθούν ώστε να αξιολογηθούν οι αρμόδιοι, οι αναγκαίοι συντελεστές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την ε, σύνταξη της τελικής έκθεσης αξιολόγησης υπάρχει μια αξιολόγηση η οποία θα πρέπει να γίνεται και δεν είναι κάτι το αυτόματο αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ. Θα σας δώσουμε και μια ένα αντίγραφο του κανονισμού 1467 και θα τα βρείτε όλα εκεί. Ο Μάρκο Βάλι δεν είναι εδώ. Ο κύριο Χόκμα είναι εδώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπερές αρχίζει να κουράζεται τώρα που θα, θα θέσω εγώ τι ερωτήσει μου. Είναι αργά πια. Και μερικέ φορέ, όσο περισσότερο ακού κάποιον, ε, τόσο περισσότερο μπερδεύεσαι. Έχω την αίσθηση ότι προσπαθείτε να τετραγωνίσετε τον κύκλο. Γιατί σε ό,τι αφορά αυτό το θετικό δημοσιονομικό προσανατολισμό και την ευελιξία, από τη μία πλευρά μα λέτε ότι πρέπει να υπάρχει ευθυγράμμιση με το σύμφωνο σταθερότητα. Δηλαδή, αυτοί που έχουν περισσότερο δημοσιονομικό θετικό προσανατολισμό, ε, θα είναι πιο σύμμορφοι. Αλλά τότε δεν χρειάζεται, ας πούμε, περισσότερη πολιτική δράση. Και από την άλλη, αυτοί που συμμορφούνται με τους κανόνες του ελλείμματος έχουν πρόβλημα με το χρέος, γιατί θα πρέπει να μειώσουν και το χρέος. Παράλληλα, είναι εντυπωσιακό ότι παρά τα πολύ χαμηλά επιτόκια, τα κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν να μειώσουν τα ελλείμματα από όσο τα μείωσαν. Παρά το πολύ χαμηλό κόστος των επιτοκίων. Τι σημαίνει αυτό αυτό, αυτός ο θετικός δημοσιονομικός προσανατολισμός. Δηλαδή, σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη δεν συμμορφούνται με τους κανόνες. Και αυτοί που δεν συμμορφούνται μπορούν να συνεχίσουν να μην συμμορφούνται. Μην ξεχνάμε ότι επιτρέπεται σε διάφορα κράτη-μέλη να μην ε, συμμορφούνται με τους κανόνες χωρίς να παίρνετε καμία δράση. Ή θεωρείτε ότι ηγηκε η ώρα να δράσουμε για τη μείωση του ελλείμματος, γιατί έχουμε μια ιστορική ευκαιρία με αυτά τα πολύ χαμηλά επιτόκια. Αν δεν μπορείς να μειώσεις το ε, έλλειμμα τώρα, θα είναι όλο και πιο δύσκολο. Όταν φτάσουν σε φυσιολογικά επίπεδα, επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα τα επιτόκια να το κάνεις. Και επίσης, σε ό,τι αφορά το, την ποιότητα των ε, προπολογισμών, δεν κατάλαβα ποτέ γιατί οι πιο σημαντικές ε, δαπάνες θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από το 103,1%. Γιατί δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέχρι από το, ας πούμε, από το 100% ας πούμε, δηλαδή σκελισμένους προσανατολισμούς. Γιατί πρέπει να περάσουμε πέρα από το 103% ε, Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί δηλαδή θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το 103% του συμφώνου σταθερότητα, στο ανώτατο δηλαδή όριο, ενώ ούτω ή άλλω οι επενδύσει έρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Και συγγνώμη για αυτήν την ερώτηση δηλαδή, αλλά είναι τόσο αργά που πια κανεί τέτοιου τύπου ερωτήσει κάνει. Yes, it's uh, Ναι, μάλλον ακριβώ είναι μια νυχτερινή ερώτηση αυτή. Και όμω είναι πολύ σκόπιμη, πολύ κέρια. Καταρχά, δεν επιτρέπουμε καμία χώρα να ξεφύγει από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το τονίζω αυτό. Όταν η Κομισιόν αυτή ανέλαβε τα καθήκοντά της, ήταν Νοέμβριος και αμέσως ετοιμάσαμε μία ανακοίνωση για την ε, ευελιξία που υιοθετήθηκε στις 13 Ιανουαρίου του 2015. Και αυτή η ανακοίνωση δεν μιλάει για αλλαγή του συμφώνου, για μη σεβάσμα του συμφώνου, αλλά απλώς εξετάζει τις ευελιξίες που μπορούν να συμπεριληφθούν και συμπεριλαμβάνονται στο σύμφωνο. Αυτές οι ευελιξίες χρησιμοποιούνταν και πριν. Απλώς δεν ε, είχαν απεικονιστεί σωστά με θεωρητικό τρόπο και πρακτικό τελικά τρόπο. Η Κομισιόν θέλει απλώ λοιπόν να σεβαστούμε το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Και ούτε ο Βαλντή, ούτε εγώ, ούτε οι συνάδελφοι σε καμία περίπτωση θα δεχόντουσαν μία απόφαση η οποία να εκφεύγει των κανόνων γενικά. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να πω. Τώρα, όταν θεωρούμε ότι αυτέ οι ευελιξίε είναι υπερβολικέ, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κτλ., αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που τι κάνουμε. Αλλά ποτέ δεν θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτή τη γραμμή. Δεν είναι στην εντολή μα και κάνουμε ό,τι μπορούμε, μια και είμαστε θεματοφύλακε των συνθήκων. Και σε καμία περίπτωση δεν είμαστε αυτοί που αλλάζουν τι συνθήκε. Είμαστε εδώ για να σεβαστούν όλοι του κανόνε. Δεύτερον, Τι σημαίνει το συνολικό, ο συνολικός δημοσιονομικός προσανατολισμός. Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ε, έναν, μια λογική στο σύνθεση επίπεδο. Η, η ΟΝΕ είναι σύγκληση και παρατηρούμε ότι σήμερα έχουμε υπερβολικές αποκλήσεις στην ΟΝΕ. Τρίτον, υπάρχει μια απόλυτη συνέπεια ανάμεσα αυτά που λέμε σε επίπεδο μέσων όρων και σε όσα λέμε σε επίπεδο χωρών. Αυτό που εννοούμε είναι ότι καμία υπερσημόρφωση, καμία υπόσημόρφωση. Τι σημαίνει τώρα αυτό με απλά λόγια. Αυτές οι χώρες οι οποίες δεν έχουν περιθώριο χειρισμού, δημοσιονομικού χειρισμού και που πρέπει να κάνουν εξυγίαση, θα πρέπει να προβούν στην εξυγίαση και θα πρέπει να είναι απόλυτα σύμμορφες με τους κανόνες οι υπόλοιπε όμω χώρε, οι οποίες τα πάνε υπερβολικά καλά και έχουν καλύτερα αποτελέσματα από το MTO, έχουν δημοσιονομικό περιθώριο και τους ζητάμε ευγενικά να το χρησιμοποιήσουν για επενδύσεις. Σε υποδομές. Μιλάμε και για ιδιωτικές επενδύσεις. Όταν ε, δρομολογήσαμε το σύμφωνο, το επενδυτικό του Juncker, δεν μιλούσαμε για δημόσιες επενδύσεις. Μιλούσαμε κυρίως για, για ιδιωτικές και δημόσιες όπου χρειαζόταν μόνο. Και αν δείτε το, την ισορροπία θα δείτε ότι είναι περισσότερο ιδιωτικές αυτές οι επενδύσεις. Αυτή είναι η λογική μας. Σωστό είναι ότι αν δεν ε, λάβουμε υπόψη τις, το, τα συνολικά ποσά και την συνολική ευελιξία και απλώς τους κανόνες, αυτό θα οδηγήσει σε αρνητική σε αρνητικό δημοσιονομικό προσανατολισμό ή δημοσιονομικό προσανατολισμό ύφεση. Αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Βλέπουμε βέβαια μια, μια ανάκαμψη, τη βλέπουμε, είναι πολύ αδύνατη, αλλά υπάρχει. Ευχαριστώ, Άλφερτ Σάντ. Ευχαριστώ. Όλοι εδώ είμαστε δημοκράτες πολιτικοί. Αυτό θα πει ότι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί για αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι όταν ε, οι άνθρωποι ψηφίζουν στι εκλογέ και τα ψηφίσματα. αυτό που μας λένε όλοι τώρα με τα αποτελέσματα είναι ότι δεν θέλουν άλλο το ίδιο. Ε, οι κανόνες του ΑΕΠ όπως εφαρμόζονται τόσο αυστηρά δεν δίνουν αποτέλεσμα. Είναι πολύ αυστηροί για να μπορέσουν να τους παρακολουθήσουν οι κανονικοί πολίτες και δεν ε, είναι εύληπτοι. Εδώ λοιπόν θα θέλαμε να δούμε κατά πόσο αυτά που εσεί υποστηρίζετε ότι είναι σωστά και δίκαια μπορούν να τα δεχτούν οι ψηφοφόροι, γιατί δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά και δεν αντιμετωπίζουμε τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα. Ιδίω λόγω των μακροοικονομικών χαμηλών επιδόσεων των προηγούμενων όμω επιπέδων είναι η πραγματικότητα. Για την πολιτική αστάθεια στην Πορτογαλία και την Ισπανία. Για άλλε ευρωπαϊκέ χώρε όπου παρατήθηκαν δύο πρωθυπουργοί και όπου ο πρόεδρο ε, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πολιτική. Οι λαϊκιστέ, για να μην πω βάρβαροι, είναι στο προσκήνιο. Οι πολιτικοί τι κάνουμε. Είσαστε εσεί ικανοποιημένοι με αυτό το αποτέλεσμα. Δεν νομίζετε ότι χρειάζεται να ξαναδούμε τι προτεραιότητέ μα. Δεν αισθάνεστε ότι είναι σαν να πηγαίνουμε ολοταχώ στο Τετανικό ε, κόντρα στο παγόβουνο. Δεν είναι τόσο προηγμένα και εξελιγμένα και περίπλοκα τελικά αυτά τα εργαλεία που έχετε προβλέψει. Ε, κάτι ήδη εκθέσαμε προηγούμενα στην αρχή από αρχή της συζήτησης πράγματι πρέπει να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες των πολιτών αυτό που αναμένουν οι πολίτες μας είναι ότι και σε σχέση με τα οικονομικά μεγέθη που συζητούμε θα αντανακλώνται σε σχέση με την πραγματική βελτίωση στη ζωή τους και στα εισοδήματά τους με άλλα λόγια δηλαδή πρέπει η οικονομική ανάπτυξη να γίνει πιο ολοκληρωμένη, ευρύτερη και γι' αυτό τονίσαμε ότι τα κοινωνικά θέματα και τα θέματα απασχόλησης στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έναντι άλλων ετών θέτουμε μεγαλύτερη έμφαση όσον αφορά την υπέρβαση των ανισοτήτων σε αυτή τη φάση τώρα διότι αυτό είναι κάτι που μεταξύ άλλων στοιχείων δημιουργεί αυτή την απογοήτευση στους πολίτες μας και δημιουργεί και αυτή την μάστιγα λαϊκισμού που προκαλείται από αυτή την κατάσταση και πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Είναι απόλυτα ορθό λοιπόν αυτό. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες των πολιτών μας και να εξεύρουμε τις απαντήσεις εκείνες που μπορούν να ικανοποιήσουν τους πολίτες αυτούς, τους Ευρωπαίους πολίτες και δεν είναι δυνατόν να υπαρκεστεί κανείς με λαϊκιστικές απαντήσεις και αντιδράσεις σε σχέση με την ανάπτυξη, της οικονομικής πολιτικής, τη δημοσιονομική πολιτική που ακολουθούμε που πρέπει να διέπεται από μια αηφορία. Διαφορετικά δεν θα έχει καμία χρονική διάρκεια, θα αποτύχει και θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα. Είμαστε μια πολιτική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είμαστε πολιτικά αντικοί. Και γι' αυτό πρέπει να προσθέσουμε στα θέματα ανάκαμψης το αν χρειαζόμαστε περισσότερες ή λιγότερες ε, δράσεις όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Νομισματική ε, Ένωση. Και η απάντηση είναι αν θέλουμε να δημιουργήσουμε τη σύγκληση πρέπει να δημιουργήσουμε σε ένα ευρύτερο, να δράσουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Γι' αυτό θα υπάρξει το λευκό βιβλίο, η λευκή Βίβλωσα από πλευράς μας σχετικά. Το πρόβλημα δεν είναι ότι η ίδια η Ευρωζώνη, όσα Ευρωζώνη δημιουργεί ύφεση, αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν δίνουν το πλήρες αποτέλεσμα, δεν δημιουργούν την μεγαλύτερη αποδοτικότητα από αυτή τη Ευρωζώνη. Σας ευχαριστούμε πολύ Βάλτης Ντομπρόφσκης και ε, Πιε για αυτή την πολύ αργά στο χρονικό ε, πλαίσιο ε, παρέμβασή σας στο διάλογο αυτό. Κλείνει ο διάλογος μας αυτός. Ο επόμενος διάλογος θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο, 12 Ιανουαρίου. Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά. Γεια σας.